Good morning, everyone. If there are no objections for today's agenda, then can consider uh, adopted without modifications. Καλημέρα σας. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις στην ημερήσια διάταξη, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Την 3η 24 Απριλίου από 3 ώρα το απόγευμα η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών διοργανώνει η επιτροπη προπολογισμών δημόσια ακροασή με θέμα τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και την Συμφωνία Κλίματος των Παρισίων. Ο στόχος είναι να αξιολογήσουμε τη συμβατότητα του ε, παρόντος και των μελλοντικών προπολογισμών της Ένωση με τη Συμφωνία του Παρισιού και να δούμε κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ε, και έχει επιτευχθεί να διαθέτει το 20% του προπολογισμού στο κλίμα. Είστε όλοι προσκεκλημένοι λοιπόν. Δεύτερον, μετά από την απόφαση της Ολομέλειας να παραπέμψει το θέμα της μετεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και βάσει του άρθρου 69F η διαπραγματευτική ομάδα θα έχει μένα ως επικεφαλής και θα συμμετέχει ο εισηγητής, ο κύριος Λαβίας, Λαβίας συγγνώμη, και οι σκιώδεις εισηγητές. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 25 Απριλίου. Στις 17 Μαΐου ε, είχαμε προβλέψει χρόνο για μία συνεδρίαση, αποδεσμεύεται αυτός ο χρόνος και έχουμε και κάποιες ε, αλλαγές. Να ε, καλωσορίσω την Ναταλία Παπαστεργίου, η οποία ήρθε στην γραμματεία της ΕΜΒΙ από 1η Απριλίου ε, από την Επιτροπή Αναφορών. Για σήμερα υπάρχει διερμηνία σε 21 γλώσσες και ο συνήθως διατίθεται ηλεκτρονικά ο φάκελος συνεδρίασης και η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Οι συστάσει των συντονιστών έχουν διανεμηθεί ηλεκτρονικά και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις μπορούν να ε, θεωρούνται δεκτές. Θα πρέπει επίσης να σας πω για τα συμπεράσματα των τριμερών διαλόγων, καταρχάς ε, για τα κτηνιατρικά προϊόντα, ο τρίτος άτυπος τριμερής διάλογος έγινε στις 22 Μαρτίου. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκαναν διεξοδική συζήτηση για τα πολιτικά εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την προστασία της τεχνικής τεκμηρίωσης για τι διαδικτυακέ πωλήσει ε, βρέθη συμφωνία για τη νέα διατύπωση για την παρέκκληση που θα περιλαμβάνει το άρθρο 108. Η συζήτηση έγινε με επικοδομητικό πνεύμα και ο εισηγητή και η Προεδρία επιβεβαίωσαν την πρόθεσή του να συνεχίσουν για να προσπαθήσουν να υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση στη διάρκεια τη Βουλγαρική Προεδρία. Ο επόμενο ε, τριμερή διάλογο προβλέπεται για τι 19 Απριλίου. Θα είναι και ο τέταρτο. Τώρα, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από την κατανάλυση καυσίμων για νέα βαρέα οχήματα. Ο δεύτερο και τελευταίο τριμερή διάλογο οδήγησε σε μια προσωρινή συμφωνία. Μετά τον πρώτο τριμερή διάλογο, ο οποίος έγινε στις 26 Φεβρουαρίου, έγιναν δύο τεχνικές συνεδριάσεις συμφωνήθηκαν αρκετές διατάξεις και έπρεπε απλώς να επιβεβαιωθούν σε πολιτικό επίπεδο. Οι δύο συνομοθέτες λοιπόν επέδειξαν μια κάποια ευελιξία, προσαρμόστηκαν λίγο στις θέσεις τους και έτσι καταλήξαμε σε συμφωνία για τις υπόλοιπες διατάξεις, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν διοικητικά πρόστιμα, κάποιες παραμέτρους παρακολούθησης, ε, διαφάνεια των δεδομένων, ε, τιμές ε, ε, φάσμα τιμών για την ποιότητα του αέρα και ε, πράξεις κατεξουσιοδότης και εκτελεστικές πράξεις. Η συμφωνία θα ε, υποβληθεί στην Κορεπέρ για έγκριση και κατά πάσα πιθανότητα θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Επιτροπή ΕΜΒΗ στις 25 και 26 Απριλίου. Και τώρα περνάμε στα θέματα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Ξεκινάμε για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς Ευρωπαίους ε, προϊόντα τα οποία είναι διαφορετικής ποιότητας στην ενιαία αγορά. Η συντάκτρια είναι η κυρία Μπόρζαν και σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο γνωμοδότησης. Να δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στην κυρία Μπόρζαν για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής της. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, οι εκθέσει Σέμικο και Άγκρη έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί, όπως γνωρίζετε, και έχουμε και αρμοδιότητα ό,τι αφορά τα τρόφιμα. Ε, η πρώτη εκδοχή της έκθεσης βασίζεται στις αρχικές, ε, στην αρχική συνεδρίαση των ευκαιοδών συγητών Όλοι και οι οδησηγητέ εξέφρασαν την προθυμία του ε, να εργαστούν σε επικοδομητικό πνεύμα και οι θέσει μα είναι αρκετά ε, συναφεί. Η έκθεση παραπέμπει σε μελέτε που έχουν διεξαχθεί σε ορισμένα κρατημέλη και εγώ προσωπικά εκπώνησα μια τέτοια μελέτη στην Κροατία σε συνεργασία ε, με τον αρμόδιο φορέα στη χώρα μου και πραγματικά προκαλούν σοκ ε, τα αποτελέσματα. Το, τα τρόφιμα για παιδιά, για παράδειγμα στην Κροατία, είναι λιγότερο ε, υγιεινά από ό,τι στην Γερμανία. Ε, υπάρχουν ε, λουκάνικα, βιέννης, τα οποία δεν έχουν καθόλου κρέας στην Κροατία. Και αυτό μπορεί να ζημιώσει την ανθρώπινη υγεία μακροπρόθεσμα. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα νέα κράτη-μέλη, βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αρνητικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα ε, που προορίζονται για ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, όπως οι βρεφικές τροφές και το καθεξής. Επίσης, οι καταναλωτές δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα αυτά, δεν είναι ενημερωμένοι και δεν ενημερώνονται και από τις ε, ετικέτες. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι η ίδια η σύσταση του τροφίμου. Χαιρετίζω το πιλωτικό έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα ε, συμπεριλαμβάνει δοκιμές ε, σε τρόφιμα και μη, ε, βάσει μιας μεθοδολογίας. Περιμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Χαίρομαι επίση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση σε ένα φόρουμ υψηλού για ε, την καλύτερη λειτουργία τη ε, επιστημιστική αλυσίδα. Λυπάμαι από την άλλη που οι οδηγίες της Επιτροπής οι κατευθύνσει δηλαδή που έχει δώσει δεν είναι αρκετά φιλόδοξε και δεν ε, ενθαρρύνουν και δεν ενδυναμώνουν τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό επίπεδο. Δεν ε, ε, μπορούμε να εξαρτώμεθα από τη βούληση των παραγωγών για την αλλαγή των επιχειρηματικών πρακτικών τους και ότι δηλαδή εκείνοι θα αλλάξουν την σύσταση των τροφίμων τους. Υπάρχουν βέβαια κάποια θετικά παραδείγματα για παράδειγμα, η εταιρεία Hippo το έκανε αυτό στην Κροατία, όμως ε, και πάλι ε, δεν γίνεται να το αφήσουμε στην καλή βούληση των παραγωγών. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναφορά στις ε, επιθυμίες και προτιμήσεις των καταναλωτών δεν γίνεται να χρησιμοποιείται ως ε, πρόσχημα ε, για την, που θα αιτιολογεί δηλαδή την ε, διάθεση στην αγορά προϊόντων που δεν είναι αρκετά ποιοτικά. Θέλουμε να δώσουμε τα απαραίτητα εχέγγυα στους καταναλωτές, να τους δίνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ποιότητα ή την, την τροποποίηση της σύστασης μιας τροφής. Χθες ακούσαμε από την Επιτροπή ότι τα προϊόντα διαφορετική ποιότητα θα καταργηθούν, θα απαγορευθούν, Θα προτιμούσα αυτή η απαγόρευση να συμπεριληφθεί σε ένα παράρτημα για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές, τη σχετική οδηγία. Γιατί αυτό είναι που πραγματικά καταλαβαίνουν οι παραγωγοί. Εναπόκειται σε εμά να κάνουμε ό,τι πέρα από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε την ίδια ποιότητα ε, τροφίμων σε όλα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για όλους τους πολίτες μας. Λαμβάνω υπόψη και την πρόταση του ΕΛΚ. Θεωρούμε, θεωρώ ότι μπορούμε να την λάβουμε υπόψη, να την συμπεριλάβουμε. Προθεσμία τροπολογι... Ε, κατάσταση τροπολογιών 23η Απριλίου. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα στους κοιόδες. Ο κύριος Πιέτσα. Σε Πιέτσα. Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, chciałem podziękować Pani Poseł. Ευχαριστώ πολύ. Jako przedstawiciel grupy EKR deklaruję. Ως εκπρόσωπος ε, της ομάδας CCR είμαι πολύ ικανοποιημένος που το θέμα των προϊόντων διπλής ποιότητας το αντιλήφθηκαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ασχολείται η Επιτροπή μας με το θέμα αυτό διότι θεωρώ ότι πρέπει να διευκρινίσουμε πολύ καλά το όλο θέμα, όχι μόνο όσον αφορά τα τρόφιμα, αλλά και άλλα προϊόντα. Παραδείγματο χάρη χημικά προϊόντα καθαρισμού. Το σημείο 6 της γνωμοδότησης ε, λέει ότι τα προϊόντα τα οποία πολλούνται στην ενιαία αγορά θα πρέπει να διαθέτουν την ίδια σύνθεση και ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται καταλήλως για οποιαδήποτε απόκληση στη σύνθεση των προϊόντων. Η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει να είναι η ίδια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραγωγοί λένε ότι όλες αυτές οι διαφορές οφείλονται στις ε, προτιμήσεις ε, των καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο. Αυτό είναι παράλογο κατά την άποψή μου. Το σημείο 5 λέει ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως αιτιολογία για ένα προϊόν, διατίθεται προϊόντα διαφορετικής ποιότητας. Οι καταναλωτές δεν... Ε, ή μάλλον οι παραγωγοί δεν μπορεί να γνωρίζουν ε, τι προτιμήσεις έχουν οι Τσέχοι, οι Πολωνοί, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί οι καταναλωτές. Οι παραγωγοί δεν λένε βάσει ποιων στοιχείων άλλωστε ε, μπορεί κάποιος καταναλωτής να θέλει να περιλαμβάνει ένα προϊόν λιγότερο ψάρι στα η περισσοτερο φινικέλο σε καποια αλλα προιοντα και οτι ειναι διαφορετικες οι προτιμησεις στην πολωνια η στη γερμανια πολυ συχνα λοιπον τα μεσα λενε οτι η δυση θεωρεί ότι η Ανατολική Ευρώπη είναι ο σκουπιδότοπος της Ευρώπης και εκεί στέλνουν προϊόντα κατώτερης ποιότητας. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε ιδιαίτερα και όλες αυτές τις απλουστεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή του λεγόμενου προϊόντος αναφοράς, διότι συνήθως Οι παραγωγοί γνωρίζουν ε, ποιες είναι οι καλές και οι κακές ε, ε, εταιρείες, παραδείγματος χάρη. Ένας παραγωγός Χ στέλνει στην αγορά συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ κάποια άλλη παραγωγή δεν είναι τόσο καλή. Κάποια προϊόντα θεωρούνται καλά και κάποια άλλα λιγότερο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πάρα πολύ καλά τη σύνθεση, τα συστατικά των προϊόντων. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που αναφέρεται εδώ ε, η εκπόνηση μιας μεθοδολογίας και ε, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και σε τοπικό επίπεδο. Εδώ ε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι προφανής και νομίζω ότι αυτός ο ρόλος θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ισορροπημένος. Το ECR υποστηρίζει την ε, γνωμοδότηση αυτή, υποστηρίζει και τη μέθοδο και προτείνει να υπάρχει μία αναλογική πίεση προς τους παραγωγούς. Εμείς όμως κυρίως ε, κάνουμε έκκληση για προσοχή Δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες στα σχέδια της νομοθεσίας. Θα πρέπει να χρησιμεύουν για την τυποποίηση των προϊόντων και την καταπολέμηση ε, των προϊόντων διαφορετικής ποιότητας. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κ. Σκύλακ. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Μπόζαν για το σχέδιο γνωμοδοτήσεως που συνέταξε, καθώς και για την πρωτοβουλία που ανέλαβε για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως των πιο ευάλωτων ομάδων, δηλαδή αυτών που ζουν στην Ανατολική Ευρώπη και που θίγονται περισσότερο από την διαφορετική ποιότητα τροφίμων που διοχετεύονται στις αγορές τους. Πρόκειται για προϊόντα που όταν πολλούνται σε όλες τις ε, χώρες μέλη εμφανίζονται καμιά φορά να είναι διαφορετικά σε κάποιες χώρες μέλη. Με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στα τρόφιμα και σε προϊόντα σχετιζόμενα με τρόφιμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό δηλώνει ότι προωθεί την καινοτομία στην αγορά και προσφέρει ευκαιρίες και σε παραγωγούς και σε καταναλωτές. Όμως, η επιτυχία μιας συγκεκριμένη επιχείρηση και η ελκυστικότητα κάποιου προϊόντος δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα απέναντι στην προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, που αυτή είναι το αγαθό που πρέπει να διαφυλαχτεί δεν μπορούν να διαφέρουν τα προϊόντα κατά την ποιότητά τους από τη μια χώρα στην άλλη, όταν το όνομα είναι το ίδιο και η συσκευασία είναι η ίδια. Εδώ συμφωνώ απολύτως με την κυρία Μπόζαν. Το να παραπέμπουν στις προτιμήσεις των καταναλωτών είναι φιλοσικής και δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται να το επικαλούνται για να φέρνουν στην αγορά προϊόντα χαμηλής ποιότητας. Εμείς γνωρίζαμε το προβλήματα αυτό, αυτά της διπλής ή διαφορετικής ποιότητας ε, των προϊόντων και αυτά δεν περιορίζονται μόνο στο τρόφιμα αλλά και σε προϊόντα υγιεινής ή καλλιντικά. Χρειάζεται λοιπόν να φροντίσουμε να συνειδητοποιήσει το κοινό το πρόβλημα αυτό και να εφαρμόσουμε μέτρα για την σωστή τήρηση της νομοθεσίας για την εξασφάλιση ίσης ποιότητας προϊόντων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και οι πολίτες της, ε, των χωρών της Δυτικής Ευρώπης όταν ταξιδεύουν σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης για ε, επιχειρήσεις ή τουρισμό θα πρέπει και αυτοί να βρίσκουν εκεί τα ίδια προϊόντα στην ίδια ποιότητα που βρίσκουν στις χώρες τους και όχι χαμηλότερη ποιότητα. Πρόκειται λοιπόν για έναν αγώνα που θα εξασφαλίσει την ίση ποιότητα προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Εργάζομαι ως και ο και εγώ για το κείμενο αυτό και ε, θέλουμε να αναγκάσουμε τα θεσμικά όργανα να εξασφαλίσουν ίση ποιότητα για όλους τους καταναλωτές γιατί αυτό θα αποτελέσει την βάση, το κείμενο μας δηλαδή, και για άλλες γνωμοδοτές για τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, η κυρία Κονέτσνα. Ε, ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για την θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει. Έχω να πω ότι το σχέδιο γνωμοδοτήσεως περιλαμβάνει λίγο πολύ όλα όσα θα ήθελα εν τέλει να δώσει το κείμενο. Χαίρομαι που το σημαντικό αυτό θέμα γίνεται πλέον προτεραιότητα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Διότι αυτά που οι πρακτικές που εντοπίζουμε αντιβαίνουν στις ε, αρχές της ενιαίας αγοράς. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια. Ήμουν παλαιότερα ε, αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τα θέματα αυτά. Και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε τις διεκδικήσεις μας. Όμως δεν έχει λήξει το θέμα, είναι αντιθέτως πολύ επίκαιρο. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε σωστές λύσεις. Η δέσμη μέτρων που προτάθηκε χθε προωθεί κάποιες λύσεις στο πρόβλημα. Όμως οι λύσεις αυτές δεν είναι επαρκείς και δεν είναι καθολικές. Το πρόβλημα αναφέρεται μονάχα στο άρθρο 6 τη οδηγία για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Δεν είναι όμως, αναφέρεται όμω και στο μαύρο κατάλογο, στη μαύρη λίστα. Αυτό είναι λάθος, γιατί έτσι υπονομεύεται η πρόταση. Επίσης, στην ε, αιτιολογική έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει ε, να ληφθούν υπόψη κάποιε προτιμήσει καταναλωτών σε ορισμένες χώρες. Αυτή είναι μια παλαιά πρόφαση πολλών παραγωγών και είναι όμως για μας απολύτως απαράδεκτη. Πρόκειται για ψεύδος, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ούτε μου αρέσει ότι επιτρέπεται να βγαίνουν στην αγορά διαφορετικά προϊόντα με την ίδια συσκευασία. Ισχυρίζονται η παραγωγοί ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να επιτρέψουν στους καταναλωτές να αγοράσουν καλής ποιότητας προϊόντα. Αυτό είναι επίση ψεύδος και πρέπει να αποκαλυφθεί. Οι καταναλωτέ θα έχουν στα χέρια τους ωστόσο τις συλλογικέ αγωγέ που είναι ένα ισχυρό όπλο. Εάν θεωρείτε ότι θα μας επιτρέπεστε εσείς από ε, την δεξιά πλευρά του φάσματος να κάνουμε μια πρόταση και μετά θα την τορπιλήσετε όπως έγινε στην Επιτροπή Γεωργίας. Εγώ σας προειδοποιώ ότι οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης είναι πανέτοιμες να θεσπίσουν ίδια δική τους νομοθεσία. Η Ουγγαρία δήλωσε ήδη ότι συντάσσει ιδιαίτερη νομοθετική πρόταση για να αντιμετωπίσει το ζήτημα των ε, προϊόντων δύο ποιοτήτων. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική που διαθέτουμε. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν θέλουμε εμείς στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες να γίνουμε το καλάθι αχρήστων της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Άλλος, κανείς, σας παρακαλώ, από τους κοιόδης, τότε το λόγο μπορεί τα μέλη. Ο κύριος Πόρκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θαυμάσια η εργασία της κυρίας Μπόζαν. Μία μικρή τεχνική παρατήρηση. Όντω χρειάζεται μια ενιαία μεθοδολογία δοκιμασιών για την, για την ε, ποιότητα των προϊόντων. Χρειαζόμαστε όμως και μια ενιαία ερμηνεία των συμπερασμάτων, των αποτελεσμάτων ε, των δοκιμασιών αυτών. Εγώ λοιπόν θα συντάξω σχετική τροπολογία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλος, κανείς, η κυρία Μποναφέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και την συντάκτρια την κυρία Μπόρζαν που με το σχέδιο γνωμοδότησης ε, προτείνει κάποια θέματα με τα οποία συμφωνώ απόλυτα. Να έχουμε ποιότητα ε, και ασφάλεια στα προϊόντα για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Και ίσως αυτό σημαίνει καταρχώς να ε, αντιμετωπίσουμε τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές που πάντα ήταν προτεραιότητα εδώ του Κοινοβουλίου. Όμως, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προσέξουμε να μην συγχαίουμε αυτό το στόχο, ο οποίος σίγουρα είναι ευγενής, με την ε, ανάγκη να επιβάλλουμε κανόνες στην ομοθέσια, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που ε, ουσιαστικά ανοίγουν το δρόμο για ένα ενίο προϊόν στα 28 κράτη-μέλη. Διότι η διατροφική παραγωγή και η σύνθεση ενός προϊόντος με την ίδια εμπορική ονομασία μπορεί να έχει διαφορετικά ε, συστατικά, εάν ε, όμως αυτά δικαιολογούνται από άλλα αίτια. Για παράδειγμα, ο χώρος παραγωγής ή συγκεκριμένες απαιτήσει παραγωγής ή και η προέλευση των πρώτων υλών λόγω και της ε, διαθέσιμότητά τους που είναι και εποχιακή, όχι μόνο γεωγραφική. Αυτό βέβαια το λέω Χωρίς παρεξήγηση, αυτό δεν σημαίνει ότι νομιμοποιείται η διάθεση στην αγορά προϊόντων χαμηλής ποιότητας και ε, φυσικά αυτό δεν πρέπει να είναι εις βάρος της ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ θετικό λοιπόν, όπως είπε και η συγγήτρια, τα όσα έγιναν ε, μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ιδίω ε, θεωρώ ότι είναι θετικό βήμα οι κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάστηκαν πέρσι. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ανατέθηκε στο Κοινό Κέντρο ε, το καθήκον να αναπτυχθεί μια μεθοδολογία για να ελέγχεται η ποιότητα των τροφίμων, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο ε, εργαλείο ε, στα κράτη-μέλη για να γίνονται και συγκριτικές δοκιμές στα κράτη-μέλη και υπό αυτή την οπτική θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κάνει περαιτέρω προσπάθειες για να αναπτύξει μια εναρμονισμένη και συνεκτική προοπτική και για να βελτιώσει το ε, νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει. Να υπάρχει ενημέρωση των καταναλωτών και να μην ε, παραπλανώνται από αθέμητες εμπορικές πρακτικές ε, που είναι αυτές οι οποίες θέλουμε στην πραγματικότητα να καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Αυτή τη στιγμή συζητούμε μια γνωμοδότηση που στόχο έχει να εγγυηθεί ότι τα προϊόντα θα είναι της ίδιας ποιότητας παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχει και ένα βαθύτερο πολιτικό μήνυμα που υφέρπει και δεν είναι τυχαίο που η συντάκτηρα της νομοδότησης, ε, καθώς ε, επίσης και οι περισσότεροι από αυτούς που έλαβαν το λόγο, είναι από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Όταν αυτές οι χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας είπαν ότι θα, δημιουργήθηκε ο ίδιο, θα δημιουργηθεί ο ίδιος ευρωπαϊκός οίκος με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις για τους πολίτες. Εάν προσπαθήστε να εξετάσετε γιατί επιβεβαιώνεται ο ευρωσκεπτικισμός ε, στην περιοχή μας, ε, η απάντηση είναι σαφής, διότι πολύ συχνά ε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν γίναμε δεχτεί στα σαλιώνα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να ερμηνεύσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες και υπ' αυτό το πνεύμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω την κυρία Παρνάση, τον κύριο μάλλον. Άντζελο Βιέκο um, uh, από την ομάδα, τη σχετική μονάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πάρω το λόγο ξανά του ε, συναδέλφου. Θα ήθελα και καν να ευχαριστήσω την Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα την κυρία Μπόρζαν για την πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει ε, στον τομέα τη διαφορετική ε, διαφορά ποιότητα στα τρόφιμα. Νομίζω ότι υπάρχει ευρύτερη στήριξη και για τόσο έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτόν τον τομέα. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εργαστεί με μεγάλη προσήλωση σε αυτό το τομέα από την αρχή για τη διόρθωση του ζητήματος. Ο πρόεδρος μας κ. Γιούγκερ καθώς και η Επίτροπος Αγιούροβα ξεκαθάρισαν ε, πολλές φορές και πιο συγκεκριμένα και πέρσι στην ομιλία για την κατάσταση ε, της Ένωσης πέρασε τον Σεπτέμβριο ότι είναι απαράδεκτο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συγκεκριμένε ε, χώρε, να διατίθεται στην αγορά ε, προϊόντα χαμηλότερη ποιότητα από τι άλλε, παρότι η συσκευασία είναι ίδια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ιεραρχήσει ω μία από τι βασικέ τη πολιτικέ προτεραιότητε αυτό το θέμα στην θητεία αυτή. Τώρα, η προσήλωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταφράζεται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Και να επενθυμίσω εν συντομία ε, τις ενέργειες που έχουμε αναλάβει σε αυτό το πλαίσιο. Πρώτον, διάλογος με τον κλάδο. Από την ε, αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί σημαντικό ε, να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφέρομενα μέρη και ιδίως ο κλάδος για να αποτρέψουμε τέτοιου είδους πρακτικές. Και αυτό έγινε στο πλαίσιο του υψηλότερο δυνατού φόρουμ που έχουμε για τέτοια πράγματα, το ε, φόρουμ υψηλού επίπεδου για την καλύτερη λειτουργία της επιστημιστική αλυσίδα. Μετά, χρηματοδότηση. Χρηματοδοτούμε και εκπονούμε ε, μελέτες ε, με μια μεθοδολογία την οποία παρουσιάζουμε και θα είναι έτοιμη, προετοιμάζουμε και θα είναι έτοιμη στα τέλη του μήνα και μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα γίνουν και πραγματικές δοκιμές ε, στα κράτη-μέλη. Κατευθυντήρες γραμμές έχουν υιοθετηθεί για να γίνεται καλή χρήση των ε, υφιστάμενων κανόνων. Και αυτό έγινε πέρσι το Σεπτέμβρη. Και έχουμε δώσει και χρηματοδότηση προς τα κράτη-μέλη για να αναπτύξουν ε, έργα και να κάνουν δοκιμές ακριβώς για το ζήτημα της διαφοράς ποιότητας στα τρόφιμα. Το καινούριο στοιχείο σήμερα και με τα χαράς ε, ανακοινώνουμε, όπως αναφέραν και κάποια μέλη, ε, ότι χθε έγινε ένα σημαντικό βήμα, ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ε, αποτροπή των διακρίσεων στα τρόφιμα στην εστρική αγορά. Έχουμε παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πακέτο, μια νομοθετική δέσμη, ε, μέσω μια τροποποίηση τη οδηγία για τι αθέμητε εμπορικέ πρακτικέ θέλουμε να γίνει αθέμητη πρακτική η ε, ε, διάθεση στην αγορά ενό προϊόντο ω ταυτόσιμου ε, όταν ουσιαστικά διαφέρει σημαντικά σε ό,τι αφορά την σύνθεσή του σε σχέση με προϊόντα σε άλλες χώρες. Θεωρούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία αυτή η πρόταση είναι ιδιαίτερος φιλόδοξη. Πρώτον, διευρύνει τη συζήτηση που προς το παρόν αφορά μόνο τα, προϊόντα, τα, μόνο τα τρόφιμα, τη διευρύνει λοιπόν σε όλα τα προϊόντα στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Μιλούμε πλέον δηλαδή για διακρίσεις προϊόντων. Με βάση τα στοιχεία βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα προϊόντα που πλήττονται από τέτοιου είδους ε, πρακτικές. Δίνουμε λοιπόν ε, αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά την πρακτική αθέμητη, αλλά συμπεριλαμβάνουμε και διατάξεις για την βελτίωση της ε, επιβολής του νόμου σε ό,τι αφορά την ε, νομοθεσία αυτή, για να προστατεύσουμε καλύτερα τον καταναλωτή από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Πώς το κάνουμε αυτό, Πρώτον, προτείνουμε και στο νομοθετικό πακέτο οι καταναλωτές να μπορούν να προσφύγουν νομικά και μεμονωμένα όταν ε, ε, πέφτουν θύματα τέτοιου είδους πρακτικών και με οικονομική αποζημίωση και με άλλα μέσα. Μετά προτείνουμε την εισαγωγή ε, πραγματικών κυρώσεων σε όταν έχουμε παραβάσεις αυτής της νομοθεσίας καταναλωτικού δικαίου και στον τομέα της ποιότητας ε, των τροφίμων. Και αυτές μπορούν να ανέρχονται και στο 4% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αυτό το κράτος Και θέλουμε να δώσουμε και ορισμένα καλύτερα μέσα στους καταναλωτές και στις ενός καταναλωτών ε, για να προσφεύγουν σε τέτοιου είδους ε, υποθέσεις. Οπότε έχουμε και τον ίδιο στόχο δεν μπορούμε να δεχτούμε τέτοιου είδου πρακτικέ, να πολλούνται δηλαδή προϊόντα διαφορετικής ποιότητας. Και εμείς έχουμε αποδείξει ε, πόσο σημαντικό είναι για μας αυτό το ζήτημα, πόσο θέλουμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδου πρακτικές, κλείνοντας να πω ότι έχουμε μία νομοθετική πρόταση, είναι φιλόδοξη και αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουμε για να πούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι βασιζόμαστε και στην δική σα στήριξη για να περάσει από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η Πρόεδρο. σας ευχαριστώ. Θα δώσω πάλι το λόγο στην ε, κυρία Μπόζαν, αλλά πρώτα στον κύριο Τουρκάνοφ. Ορίστε. Ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να προσέλθω κυρία Πρόεδρε. Ε, είχα άλλη ανηλυμένη υποχρέωση. Μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα που συζητούμε την ε, πρόταση αυτή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για μας που εκπροσωπούμε τα συμφέροντα των πολιτών των ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή η δυτή ποιότητα υπάρχει σε χώρες όπως Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία επίσης, τη χώρα μου δηλαδή, την οποία πω εγώ, εμείς έχουμε εδώ λοιπόν πιστικά επιχειρήματα για να δεσμευτούμε για τον αγώνα αυτόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο έθεσαν και άλλοι συνάδελφοι προηγουμένω και έχω να προτείνω και να κάνω και κάποιε προτάσει για το πώ είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό της διαφορετικής ποιότητα Χαίρομαι για την ε, γνωμοδότηση. Δεν μπορούν οι προτιμήσεις των καταναλωτών να χρησιμοποιούνται ως πρόφαση για να διοχετεύονται στην αγορά προϊόντα διαφορετικής ποιότητας. Εδώ θα πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου, διότι συχνά χρησιμοποιούνται τα επιχειρήματα αυτά ως προφάσεις για αθέμητες πρακτικές. Έχω συνομιλήσει με εκπροσώπους ε, οργανώσεων των καταναλωτών αλλά και των παραγωγών και μου λένε ότι ναι, κοιτάξτε, είναι διαφορετικές οι γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών σε διάφορες χώρες μέλη. Δεν θα πρέπει να είναι όμως επιτρεπτό να είναι διαφορετική η σύνθεση επειδή έχουν διαφορετικές προτιμήσεις οι καταναλωτές. Ούτε είναι άλλωστε δυνατόν να ε, επιδεινώνεται η ποιότητα του προϊόντος για να κάνουν εξοικονομήσεις κόστους η παραγωγή. Ίσως να τα έχετε πει αυτά τα πράγματα ήδη. Γι' αυτό και ζητώ συγγνώμη που τα επαναλαμβάνω. Αλλά έχω να πω κάτι ακόμη. Το οποίο άκουσα από ρουμανική οργάνωση καταναλωτών. Γίνεται πρόταση να εισαχθούν νέοι έλεγχοι. Σύμφωνα δηλαδή, μάλλον ε, να είναι ε, εξέταση του προϊόντος δοκιμασία, επιθεώρηση. Αυτά στον τομέα ασφάλειας των τροφίμων. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ιδρυθεί ο οργανισμός, ο οποίος να αναλάβει τις αρμοδιότητες αυτές, να ελέγχει δηλαδή την ποιότητα των προϊόντων, εφόσον υπάρχει σχετική υποψία διαφορετικής ποιότητας, Υπάρχουν πολλές προτάσεις. Ολοκληρώνω τώρα. Υπάρχει χρόνος ακόμη για να τοποθετηθούν, ε, για να ε, καταθούν τροπολογίες. Εγώ οπωσδήποτε θα υποβάλω τροπολογίες. Ελπίζω, θε, ότι η γνωμοδότηση της κυρίας θα αποτελέσει ισχυρό μήνυμα προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται να λάβει αποφάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την... Μάλλον να δώσουμε το λόγο στην κυρία Παζόνη για τα καταπληκτικά της σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους συναδέλφους και τους ασκιώδεις και τους υπόλοιπους ε, προβουλευτές που έχουν συμβάλει στη συζήτηση. Συμφωνώ με τα περισσότερα των σχολείων σας, ιδίως με τα όσα είπε η κυρία Κονέτσνα. Ο κύριος Καρλέτς επίσης είπε ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε και στους πολίτες της Δυτικής Ευρώπης. Όσοι από εμάς ε, νιώθουμε ότι μας επηρεάζει αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να εξηγήσουμε στους πολίτες περί τίνος πρόκειται. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη μεθοδολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και περιμένω ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Θεωρώ επίσης ότι αυτός ο διαχωρισμός μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης ως προς την ποιότητα τροφίμων προϊόντων μάλλον, δεν είναι πολύ θετική εικόνα από τη μελέτη που κάναμε στην Κροατία, όπως είπα και στην αρχή της συνάντησής μας, ε, προέκυψε ότι τα γενέζικα λουκάνικα στην κροατική αγορά δεν έχουν καθόλου κρέας, ενώ είναι πάνω από 6% στην ε, ε, Γερμανία. Ενώ αυτό το προϊόν διατήθηκε διατίθεται και στην Ιταλική αγορά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και οι Ιταλοί καταναλωτές πλήττονται από αυτού του είδους την πρακτική. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε τα αποτελέσματα ε, προκειμένου να έχουμε τη στήριξη των βουλευτών και από την Ανατολή και από τη Δύση και να είναι όλοι οι ευρωβουλευτές ενωμένοι γιατί πρόκειται για τα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων καταναλωτών όπως ε, εγγράφεται ε, στα κείμενά μας. Και συμφωνώ και εγώ ότι αυτή η πρακτική είναι πραγματικά παράδεκτη. Ο κύριος Γιούνκερ επίσης αναγνώρισε αυτό το πρόβλημα γιατί εάν δεν το είχε πράξει δεν θα είχε αφιερώσει το σημαντικό τμήμα της ε, ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης αναφέροντας ότι πρέπει να σκεφτόμαστε την Ένωση ως σύνολο και όχι με γεωγραφικούς προσδιορισμούς. Για τα όσα είπε η κυρία Μποναφέ, ότι υπάρχουν προτιμήσεις των καταναλωτών. Κατανοώ ότι οι παραγωγοί επιθυμούν να τροποποιήσουν τα προϊόντα τους με βάση αυτές τις προτιμήσεις όμως. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ε, στις σοκολάτες που διατίθενται στην Ανατολική Ευρώπη χρησιμοποιούνται υποκατάστατα ορισμένων ε, ε, ουσιών αντί για την πραγματική ουσία. Συμφωνώ και με τον εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Είπα και εγώ εισαγωγικά ότι θα λάβουμε υπόψη τις τροπολογίες σας για τις για τους επιτόπιους ελέγχους. Νομίζω ότι πραγματικά αυτό είναι απαραίτητο. Πρέπει λοιπόν να θέσουμε τις βάσεις ε, για νέους ε, κανόνες που θα μας επιτρέψουν να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα ε, και θα εξηγήσουμε σε όλους τους φορείς ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους ε, πολίτες μας και να υπενθυμίσω ότι χωρίς τους πολίτες και χωρίς εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχε εντοπίσει αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους που ε, επισημάνατε αυτό το ζήτημα. Όπως ήδη ανέφερε η συγγήτρια, μέχρι τις 23 Απριλίου μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Πιθανώς να ψηφίσουμε στην ΕΜΒΗ στις 20-21 Ιουνίου. Φτάνουμε στο τέλος αυτού του σημείου. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο, ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, πιθανές περαιτέρω, ε, πιθανό περαιτέρω περιορισμό για την χρήση των νέων νοικοτινοειδών. Θα ξεκινήσουμε με την Επιτροπή και μετά δώσουμε το λόγο στα μέλη μας. Ο κύριος Κλάους Βέρεντ είναι μαζί μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ε, ε, Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Το θέμα αυτό, το οποίο προτείνεται να συζητήσουμε σήμερα, έχει αρκετά στο ιστορικό του. Ε, πριν από μια δεκαετία ε, περίπου διαπιστώθηκε ότι κάποια φυτοφάρμακα τα οποία περιλαμβάνουν ε, νεονικοτινοειδή αποτελούν πολύ σημαντικό κίνδυνο, ε, κίνδυνο για τις μέλισσες. Έτσι το 2013 ε, απαγορεύτηκαν τρεις νεονικοτινοειδείς ουσίες και αυτές οι ουσίες ε, δημιουργούν προβλήματα, η κλωριαδίνη, η θυμεδοξίνη και η μαδοκλοπρή. και αυτές ε, απογορεύτηκαν σε περιοχές ε, ε και σε θερμοκήπια τα οποία και είδη τα οποία χρησιμοποιούνται πριν από τη σπορά. Ε, αποφασίστηκε ότι θα γίνεται έρευνα για όλες τις νέες ε, επιστημονικές πληροφορίες πριν τεθεί σε εφαρμογή, ε, δηλαδή μέχρι το Μάιο του 2015 ο νέος κανονισμός. Ε, οι παραγωγοί υπέβαλαν τα στοιχεία συμμόρφωσης ε, στην Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο του 2016 δημοσίευσε τα συμπεράσματά της. Βάσει αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και για τις τρεις στοιχείες ε, ουσίες, ε, ακόμα και αυτά τα οποία είναι ακόμα εγκεκριμένα και ξερούνται δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή. Επομένως, ε, περιορίστηκε περαιτέρω η χρήση αυτών των ουσιών και συζητήθηκε προτάσεις με τα κράτη-μέλη από τον Οκτώβριο του 2017 και μάλιστα έγινε μια συζήτηση και για αυτές τις προτάσεις πέρσι τον Ιούνιο εδώ στην Επιτροπή σας όταν υπήρχαν αρκετές ε, ενστάσεις ε, οι οποίες τελικά δεν εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Μάιο του 2017 Ανακοινώσαμε το σχέδιο κανονισμών επισήμω ε, στον ΠΟΕ βάσει τη συμφωνία για προσκόμματα στο εμπόριο. Ε, Επομένω, υπάρχει υποχρέωση για να δίνεται η δυνατότητα σε τρίτε χώρε για να σχολιάσουν τι προθέσει μα. Και αυτό ξεκίνησε και μία περίοδο 60 ημερών για να ληφθούν αυτά τα σχόλια, η οποία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Μετά προτείναμε και προβλέπαμε να ψηφίσουμε το σχέδιο κανονισμών στην Αρμόδια Επιτροπή ε, για τα φυτά ε, το 2017, αλλά πολλά κράτη-μέλη ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιμένει τα αποτελέσματα της γενικότερης αναθεώρησης που έκανε ο ΕΦΣΑ ε, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Και αυτή η αναθεώρηση είχε ξεκινήσει εγκαίρως, ε, ζητήθηκε από την ΕΦΣΑ να ε, ε, κάνει ανοιχτό διαγωνισμό για συλλογή στοιχείων που έγινε από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τον ΕΦΣΑ να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που υπευλήθησαν καθώς επίση και όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμε από τη βιβλιογραφία. Αυτό ο ανοιχτός διαγωνισμός είχε ως αποτέλεσμα να υποβληθούν πάρα πολλά στοιχεία στον ΕΦΣΑ και χρειάστηκε πολύ χρόνος για να γίνει η αξιολόγηση που του είχε ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τελικά δημοσιεύθηκαν οι εκθέσεις στις 28 Φεβρουαρίου του τρέχοντος και ε, σε μεγάλο βαθμό ο ΕΦΣΕ επιβεβαίωσε σε αυτές τις εκθέσεις ότι η περαιτέρω χρήση αυτών των τριών ουσιών αποτελεί κίνδυνο για τις ε, άγριες μέλισσες και για τις ε, μέλισσες που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομεία και γενικότερα ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτός ο κίνδυνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν διατηρεί αυτούς τα σχέδια κανονισμών που θέλει να απαγορεύσουν όλες τις χρήσεις αυτών των ουσιών και ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να ψηφίσουν τις προτάσεις στη μόνιμη επιτροπή τώρα στις 27 Απριλίου. Και αυτά λοιπόν είναι αυτά τα οποία μπορούμε να πούμε εν είδη εισαγωγή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπέρντ. Τώρα, οι συνάδελφοί μου προσκαλούνται να λάβουν τον λόγο. Ορισμένοι ήδη έχουν εγγραφεί. Ο κύριος Φλόρεντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο ίδιος συμβατικός ε, γεωργός και χρησιμοποιώ πολλά συμβατικά οκτώνα αλλά για τα νέο νοικοτινοειδή έχω πολλές αμφιβολίες. Δεν είναι κάτι το οποίο το ψεκάζεται πάνω στα φυτά, ανακατεύεται με τους σπόρους και έχει μετά μια ε, διάρκεια ε, ισχύω από ε, μέχρι χίλιες ημέρες. Έχει, έχω λοιπόν την παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο το έδαφος στο μέλλον και όχι το νερό. Συμβολικά, εάν από πάνω ρίξετε κάτι στο έδαφος και μετά δεν βρίσκεται πλέον τίποτα, ε, κάπου έχει μείνει μέσα στο έδαφος. Κάποιο από αυτό θα το επεξεργαστούν οι μικροοργανισμοί, αλλά το έδαφος είναι το κλειδί για τη μελλοντική προστασία των φυτών. Ας το λάβει υπόψη της αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πάντως ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κάτι που με ενδιαφέρει επίσης πολύ προσωπικά είναι το ερώτημα ποια επιχειρήματα έχουν οι χώρες μέλη. Θα ήθελα να μάθω και η δική μου χώρα ε, τι στάση έχει. Και ποιες αλλαγές θέλουν να επιφέρουν και πώς και πώς κρίνει τα επιχειρήματα κάποιων γεωργών που με επισκέφθηκαν και εμένα. Αν δεν έχω πλέον τα νεονικοτινοειδή, θα έχω πρόβλημα, διότι οι μικροοργανισμοί που χάνουμε διαρκώς, τους προστατεύαμε ενώ οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι που καθιστούν έφορο το ε, γεωργικό έδαφος. Πρέπει να τους προστατεύσουμε λοιπόν, σαν τα μάτια μας και γι' αυτό πρέπει να μείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκληρή και να μην ενδώσει, ακόμα και αν βρω εγώ τον πελά μου, το δέχομαι αυτό. Τα νεονικοτινοειδή είναι για την ώρα τα ε, πιο επικίνδυνα ε, βιοκτώνα συστημικού χαρακτήρα στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Φλόρεντς. Κύριος Πότς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε να ψηφίσουμε σύντομα για την απαγόρευση των νοικοτινοειδών. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Επειδή απαγορεύσει, ή μάλλον το 2013, τέθηκαν σε ισχύ από το 2013, έχουν προβλεφθεί ολόκληρες δωδεκάδες εξαιρέσεων σε πολλές χώρες μέλη και σε ορισμένες χώρες μέλη οι περιορισμοί του 2013 δεν εφαρμόστηκαν ποτέ λόγω της διαρκούς χρήσης ή κατάχρησης του συστήματος των εξαιρέσεων. Τι περιμένει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αρχίσει να προσφέρει κατά των χωρών αυτών για παραβίαση των απαγορεύσεων, των περιορισμών και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποτρέψει τις χώρες από το να χρησιμοποιήσουν τις ε, ε, εξαιρέσεις αυτές στο μέλλον, ο κ. Στάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πολύ ενδελεχή αυτή παρουσίαση για τα όσα συνέβησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ευχαριστώ επίσης για το γεγονό που ανακοινώνουν, ότι ανακοινώνουν ότι όντως θα γίνει η ε, ψηφοφορία στις 27 Απριλίου στη Διαρκή Επιτροπή. Έχω μια σειρά ερωτήματα, όπως ανέφερε ο κύριος Φλόρενς. υπάρχει ο κλάδο των ζαχαροτέφλων που ασκεί τεράστιε πιέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα να ρωτήσω, μήπω ε, θα επιτρέψει την χρήση των νεονικοτονειδών στον κλάδο αυτών. Συμφωνεί η Επιτροπή ότι η χρήση των ουσιών αυτών στα ζαχαρότευτλα δεν ε, δημιουργεί κανένα, δεν ενέχει κανένα κίνδυνο παρά την γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Θα ήθελα λοιπόν μια διακρίνηση προς αυτό. Δεύτερον, ο κύριος Πότς το έθεσε πολύ κομψά. Υπάρχουν πάρα πολλές παρεκκλήσεις, οι οποίες εκχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ε, των κρατών μελών. Ε, κάπου διάβασα είναι πάνω από χίλιες τα τελευταία χρόνια. Και μπορούμε ουσιαστικά να πούμε ότι ε, με την εκχώρηση όλων αυτών των παρεκκλήσεων μπορεί κανείς να πει ότι πλέον παρακάμπτεται αυτή η απαγόρευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να επιτρέπει αυτές τις παρεκκλήσεις, γνωρίζοντας ότι ουσιαστικά έτσι παρακάμπτεται η απαγόρευση. Τρίτον, είναι όλο αυτό το ζήτημα των θερμοκηπίων. Εκεί επιτρέπεται η χρήση των νέων οικοτινοειδών. Όμως, ε, διαβάζω και τα άρθρα που αναφέρεται ότι η χρήση των νέων οικοτινοειδών και στα θερμοκήπια ε, ουσιαστικά επηρεάζει, ενδεχομένως μολύνει και τον υδροφόρο ορίζοντα στην περιοχή αυτή. Ε, η ΕΦΣΑ το έχει μελετήσει. Υπάρχει όντως ε, πιθανός κίνδυνος. Θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό. Και τέλος, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει ψηφοφορία στις 27 Απριλίου στη Διαρκή Επιτροπή έχουμε μια μερική εικόνα μόνο σε ό,τι αφορά την στάση των κρατομελών. Ο κύριος Φλόρενς είπε ότι θα ήθελε να γνωρίζει την στάση της Γερμανίας, αλλά νομίζω ότι ε, στο πολιτικό του κόμμα είναι μέλος της πλειοψηφίας, οπότε σίγουρα μπορεί να το μάθει αν θέλει με τις επαφές ε, που έχει στο ιστορικό του κομματός του. Το ερώτημά μου προς την Κομισιόν. Αν δεν υπάρχει ε, περίπτωση ειδική πλειοψηφία στη Διαρκή Επιτροπή, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προχωρήσει παρόλα αυτά. Θα επιδείξει αρκετό θάρρο, ούτω ώστε ακόμα και αν δεν υπάρξει ειδική πλειοψηφία, να λάβει μία οριστική απόφαση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σέτεμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση. Έχω κι εγώ μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, ε, στον 1107 για την ε, προστασία των φυτών ξεκαθαρίζεται ότι πρέπει να υπάρχει κίνδυνος ε, για είδη που δεν στοχεύονται. Όμως γιατί μιλούμε μόνο για τις μέλισσε και όχι για άλλου, και για άλλους οργανισμούς, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, ποιε είναι οι επιπτώσεις ε, της ε, παραμονής αυτής της ουσίας, είτε στο έδαφος είτε στο νερό. ήθελα να μας το πείτε αυτό. είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία εύρωστη ε, επιστημονική γνωμοδότηση ως προς αυτό. Δεν πρέπει να, γίνουμε, να κάνουμε εδώ συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για να δούμε κατά πόσο είναι επικίνδυνες αυτές οι ουσίες ή, ή όχι. Όμως, σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία διοδότησης για τα, ε, για, τα προϊόντα φυτοπροστασίας, πολύ καλά, όμως ε, υπάρχουν και επιπτώσεις αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ουσίες που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, αυτήν την εβδομάδα στις κάτω χώρες υπήρξε μια μελέτη της ε, Ολλανδικής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων ότι οι επιπτώσει τη επιμέρου καλλιέργεια μπορεί να είναι τεράστιε αν απαγορεύσουμε τη χρήση των νέων οικοτενοειδών και μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο ο κίνδυνο για το περιβάλλον αν τις απαγορεύσουμε, γιατί πρέπει να έχουμε εναλλακτικέ λύσεις. Θα ήθελα να κάνουμε λοιπόν και αυτή τη συζήτηση. Πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να υπάρξει και λύση, όμως πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αν δεν συνεχίσουμε την αδειοδότηση των ουσιών αυτών, θα βρούμε μια άλλη λύση που δεν θα ε, ζημιώνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ε, θέτω αυτό το ερώτημα εξ ονόματο τη κυρία Δελανό. Την 1η Μαρτίου υπέβαλα στην Ολομέλη μια τροπολογία στην ε, έκθεση τη πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου για το μέλλον τη μελισσοκομεία, ε, στην οποία συνυπέγραψαν 75 συνάδελφοι. Δυστυχώ απερίφθη η τροπολογία. Εκεί ζητούσαμε την πλήρη απαγόρευση, χωρί καμία καθυστέρηση, όλων των κατανοητών στα ριζανιοκτώνα, καθώ ε, πλήττουν το κεντρικό νευρικό σύστημα των μελισσών και σκοτώνουν εκατομμύρια μέλισσε. Αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι επιζήμια η χρήση στα θερμοκήπια. Χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα για την ε, παράταση τη γενική απαγόρευση, όμω με ε, βάση τι νέες μελέτες, αποδεικνύεται ότι αυτά τα ε, ζανιοκτώνα παραμένουν στον υδροφόρο ριζονταϊκά, στο έδαφο για πολλά χρόνια και αποτελούν πραγματικό κίνδυνο για την βιοπικιλότητα. Ερωτώ λοιπόν γιατί σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός κίνδυνο στη χρήση των ουσιών αυτών στα θερμοκήπια. Γιατί δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. κάποιο άλλο. Η κυρία Κιούζο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η ιστορία των ε, ε, βασίζεται σε όλα αυτά που συζητούμε εδώ. Χρειαζόμαστε σοβαρές ε, και επιστημονικές ε, μελέτες και ε, όντως αποτελεί κίνδυνο για τις μέλισσες, αλλά δεν είναι μόνο τα νεονικοτινοειδή τα προβλήματα των μελισσών. Υπάρχουν ε, και άλλα προβλήματα. Όπως πολύ σωστά είπαμε, υπάρχουν συνέπειες και για τις ε, καλλιέργειες. Ε, αν αρχίζουμε να μειώνουμε το διοξίδιο του άνθρακα, ε, θα πρέπει να εξετάσουμε και τις εκπομπές των ε, αυτοκινήτων, ε, αλλά και τις εκπομπές ε, στην παραγωγή. Και πρέπει να κάνουμε τα πράγματα σοβαρά αυτή τη στιγμή, γιατί μειώσαμε τις εκπομπές στα οχήματα και τις αυξήσαμε τελικά στις παραγωγές. Πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και να λάβουμε υπόψη και τι συνέπειες θα υπάρχουν για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπόιλαν. Ευχαριστώ. Αντί να επαναλάβω τα όσα ήδη ακούστηκαν, θα ήθελα να συμφωνήσω με τα σχόλια του κυρίου Πότς. Η ε, Επιτροπή προτείνει να μειώσουμε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από τα παραθυράκια μάλλον που έχουν δημιουργηθεί από τις παρεκκλήσεις. Εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε νεονικοτινοειδή σε κάποιες ε, καλλιέργειες στα θερμοκήπια, δεν θα πατάξουμε το πρόβλημα, θα συνεχίσουν σε άλλες καλλιέργειες. Και τι θα γίνει εάν χρησιμοποιούνται στα θερμοκήπια προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα περιοριστεί η χρήση τους και δεν θα πηγαίνουν και στο ευρύτερο περιβάλλον μέσω του εδάφους και μέσω του υδροφόρου ορίζοντα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει και τι αντίκτυπο έχουν τα νεονικοτινοειδή και σε άλλα είδη και τα δύο νεονικοτινοειδή που ε, αποκλείονται από τον ε, κανονισμό του 2013. Η κυρία Κάδεμπαχ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει λίγο πολύ το ίδιο νόημα. Υπάρχουν μελέτες και έρευνες που δείχνουν ότι θα πρέπει να απαγορευτούν τα νεονικοτινοειδή με βέβαια την εξαίρεση των ε, θερμοκηπίων. Η ερώτησή μου λοιπόν αναφέρεται στο μέλλον. Χρειάζεται κάποιο monitoring, κάποια παρακολούθηση για να διαπιστώνεται εάν ίσως η χρήση σε θερμοκήπια επιβαρύνει και αυτή το περιβάλλον. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ελευθερία επιλογής εφόσον υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος κανείς? Εάν δεν υπάρχει άλλος, τότε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κ. Μπέντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλα τα μέλη σας που τοποθετήθηκαν και που γενικά ε, υποστηρίζουν τις προτάσεις μας ε, για τις επόμενες δράσεις να απαντήσω στις ερωτήσεις τώρα με τη σειρά που τέθηκαν. Κύριε Φλόρεντς, αλλά και ο κύριο Στάς, ρωτήσατε για την θέση των χωρών μελών. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τις ε, επιμέρους θέσεις των χωρών μελών που προβάλλονται στην Διερκή Επιτροπή, αλλά λίγες χώρες μέλη τον τελευταίο Μάρτιο υποστήριξαν πλήρως τις προτάσεις της Επιτροπής. Λίγες αντιτάχθηκαν και η μεγάλη πλειοψηφία δεν είχε ακόμα τελική θέση. Το βασικό θέμα που απασχόλησε την συζήτηση είναι αυτό που έθεσε και ο ε, κ. Φλόρενς, δηλαδή η παραγωγή ζαχαροτέφλων και όπως ο κ. Φλόρενς δεχθήκαμε και εμείς ε, επισκέψεις παραγωγών ζαχαροτέφλων οι οποίοι ήταν μεν φιλικοί αλλά πολύ σταθερή και η δική μας η αντίδραση ήταν φιλική αλλά σταθερή. Βεβαίω το ίδιο ακριβώς όπως με τη δική τους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται να εξετάσει εξαίρεση για την παραγωγή ζαχαροτέρθρων Απαντώ έτσι και σε μία από τις ερωτήσεις του κ. Στάς. Είναι αλήθεια ότι ο οργανισμός ΕΦΣΑ δεν έχει εντοπίσει άμεσο κίνδυνο από την χρήση των δικοτινοειδών για τα ζαχαρότευτα, αλλά όπως είπε ο κ. Φλόρεντς, η παραμονή στο έδαφος αποκαλεί, ε, αποτελεί κίνδυνο για τις επόμενες διαδοχικές ε, ε, εσοδίες που απορροφούν τα νεοδικοτινοειδή και μετά καταλήγουν αυτά στους γονιμοποιητές, δηλαδή στις μέλισσες. Άρα δεν εξετάζουμε το ενδεχόμενο εξαίρεσης για τη διαρκή χρήση για την παραγωγή ζαχαροτέφτων. Ο κ. Πότς με ρώτησε για τις ε, κατεπίγουσες αδειοδοτήσεις. Το γνωρίζει το πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε υπενθυμίσει κατ' επανάληψη στις χώρες μέλη που χορηγούν αυτές τις κατεπίγουσες εξαιρέσεις με αρκετά γενναιόδωρο τρόπο, δηλαδή καλύπτουν ολόκληρη την επικράτειά τους και πολλών ειδών παραγωγές, ότι αυτό τελικώς μας φαίνεται ότι είναι ασύμβατο με το περιεχόμενο του κανονισμού και της οδηγίας. Και ζητήσαμε από τον ΕΦΣΑ πέρσι να αξιολογήσει εάν οι χορηγούμενες κατεπίγουσες εξαιρέσεις για το 2017 από αυτούς τους κατ' επανάληψη ή τις δράστες αν είναι δικαιολογημένες. Θα λάβουμε την απόφαση του ΕΦΣΑ τον Μάιο και μετά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να απαγορεύσει στις ε, χώρες αυτές να δώσουν ξανά τέτοιου είδους εξαιρέσεις. Απαντώντας ε, και στον κύριο Στάς πάλι, θέλω να πω ότι η ευθύνη για την χορήγηση των αδειοδοτήσεων είναι καθαρά και μόνο στα χέρια των χωρών μελών δεν ε, εγκρίνει η χορηγή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από έτσι των χωρών μελών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χωρών μελών. Μπορούμε να εξετάσουμε εάν οι συνθήκες όντως πληρούνται, οι όροι δηλαδή της ε, νομοθεσίας, αλλά δεν χορηγούμε εμείς ε, επίγουσες εξαιρέσεις. Τέθηκαν ορισμένες ερωτήσεις για την διαρκή χρήση στα θερμοκήπια. Αναφέρομαι στα συμπεράσματα του ΕΦΣΑ που αποτέλεσαν την βάση για την δράση μας. Τα δε συμπεράσματα του ΕΦΣΑ στις σχετικές εκθέσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι όντως ασφαλές να χρησιμοποιούνται τα νεονικοτινοειδή στα θερμοκήπια. Θα ήθελα να τονίσω ότι βέβαια ο ορισμός των θερμοκηπίων πρέπει να είναι αυστηρός, δηλαδή μόνιμο θερμοκήπιο που σημαίνει ότι διαθέτει και σύστημα διαχείρισης που διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει διάδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και ότι τα διάφορα απόβλητα ε, γίνονται αντικείμενο της σωστής επεξεργασίας πριν να διατεθούν στο περιβάλλον. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι υπάρχει και λευκή επιταγή για την διαρκή χρήση στο μέλλον. Πάλι οι χώρες μέλη θα ε, εκδίδουν τις αδειοδοτήσεις για τα θερμοκήπια, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Και αν ανακαλύψουν τέτοιες, θα πρέπει βέβαια να ανακαλέσουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Τέθηκε μια ερώτηση επίσης σχετικά με άλλα νεονικοτινοειδή. Εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ανανεώσαμε την έγκριση του σεταμιπρίτ άλλου νεονικοτινοειδούς πάλι στην βάση των συμπερασμάτων του ΕΦΣΑ που μας διαβεβαιώνει ότι είναι χαμηλή η κίνδυνη για τις μέλισσες και άλλους γονιμοποιητές και άλλο βρίσκεται στην φάση της διαδικασίας ανανέωσης της αδειοδότησης. Η δε απόφαση θα ληφθεί προσεχώς. Η ερώτηση του κ. Χάτουμα δεν εξετάζουμε μόνο τις επιπτώσεις στις μέλισσες αλλά και σε άλλα είδη καθώς και από τα επιπτώσεις στο έδαφος και σε μικροοργανισμούς του εδάφους. Και έχουμε και σχετικό έγγραφο για το πώς πρέπει να γίνονται οι εξετάσεις αυτές. Ο κ. Χάτιμα ρώτησε επίσης εάν μας απασχολούν οι επιπτώσεις στην για την προστασία των ε, παραγωγών, της εισοδίας δηλαδή. Πρώτα, ο κανονισμός δεν προβλέπει ότι οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη όταν εγκρίνει η Επιτροπή. Αναφέρεται μοναχά στον κίνδυνο που προκύπτει από τη χρήση των νεονικοτινοειδών. Και μετά από τους περιορισμούς του 2013, το Κοινό Κέντρο Ερευνών έχει κάνει μια έρευνα για να εξετάσει τι έχει συμβεί σε σχέση με τις στρατηγικές που ακολουθούν οι γεωργοί για την προστασία των εσοδιών όταν δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον νέο νοικοτινοειδή και διαπίστωσε το κέντρο ερευνών ότι όντως οι παραγωγοί έχουν βρει κάποιες εναλλακτικές επιλογές, ανεφέρθηκε σε αυτές ο κύριος ε, ε, Φλόρενς, δηλαδή χρήση άλλων ζυζανιοκτώνων ή άλλες σταδικές διαχείρισης των ε, ζυζανίων ή άλλων επιβλαβών οργανισμών. Επομένως, οι γεωργοί μπόρεσαν να βρουν εναλλακτικές επιλογές ήδη από τότε. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό θα καταστεί δυνατόν το ίδιο και σχετικά με τις προτάσεις που καταθέτουμε τώρα. Ναι, ένα ακόμη ενημερωτικό στοιχείο σχετικά με το monitoring, το Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για την παρακολούθηση της παρουσίας των ηχνοστοιχείων ε, ε, των νοικοτινοειδών στις μέλισσες έχει γίνει πρόσκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και εκτός αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται και επί ενός ευρύτερου σχεδίου για τους ε, γονιμοποιητές όλων των ειδών και τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα όλη αυτή η συζήτηση και θα περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις στον τομέα. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι και πάλι ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, Γενική Έκθεση για την Λειτουργία του Κανονισμού ΡΙΤΣ και Αθεώρηση Ορισμένων Στοιχείων, Συμπεράσματα και Δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μία αναθεώρηση του, Ρίφιτ ε, ε, του REACH, συγγνώμη, κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα και θα συζητήσουμε σήμερα το θέμα αυτό με τον κύριο Σαντάουσκας, Διευθυντή Κυκλικής Οικονομίας και Πράσινης Ανάπτυξης στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Έχετε το λόγο λοιπόν απευθείας κύριε Σαντάουσκας. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή για μένα να με συνοδεύει και ένας συνάδελφος, ο Κάρλο Πετινέλη, από τη Γενική Διεύθυνση Grow. Και αυτό νομίζω ότι ευθύ εξ αρχή καταδεικνύει ότι πρόκειται για συλλογική εργασία, έγινε από δύο υπηρεσίε. Και αυτό είναι και ένα από του λόγου που αυτή η αναθεώρηση ήταν ιδιαίτερη. Και ήταν ιδιαίτερη και για άλλου λόγου βεβαίω. Έγινε ένα fitness check και ε, μια αξιολόγηση ε, ενός πολύ σημαντικού νομοθετήματος που θέτει και παγκόσμια πρότυπα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, καθορίζει ένα σύστημα το οποίο είναι ακόμα υποκατασκευή. Το 2006 θα θυμάστε ότι ήταν πολύ σημαντικό ορόσημο για την πολιτική χημικών στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο κανονισμός αυτός ε, ε, έθεσε την βιομηχανία ενώπιον των ευθυνών της για όλη την αλυσίδα προμηθειών και επιτάχυνε την αξιολόγηση και διαχείριση των επικίνδυνων χημικών από τις αρχές. Έγινε η πρώτη αξιολόγηση το 2010, αλλά τότε κάποια από τα κεφάλαια του κανονισμού REACH ακόμα δεν είχαν τεθεί σε εφαρμογή. Επομένως, ε, ήταν η πρώτη τα πρώτα στοιχεία αυτά τα οποία ε, εξετάσαμε. Τον περασμένο μήνα, στις 5 Μαρτίου, εγκρίθηκε η Γενική Έκθεση για την εφαρμογή του ΡΙΤΣ. Είναι η δεύτερη αναθεώρηση του ΡΙΤΣ ε, και εξέταση συγγνώμη, του ΡΙΤΣ ε, και είδαμε τις προκλήσεις μετά από 10 χρόνια εφαρμογής αυτού του κανονισμού. Όλες οι διαδικασίες του ΡΙΤΣ πλέον είναι σε εφαρμογή. Αυτό ήταν τμήμα του προγράμματος ε, εξέτασης ε, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Fitness Check, και εξετάσαμε τα βασικά στοιχεία που εξετάζει ε, το Fitness Check όταν γίνεται αυτός ο έλεγχος ε, εξετάσαμε την αναθεώρηση του REACH ε, του 2010, αλλά εξετάσαμε και άλλα στοιχεία. Είναι μια αξιολόγηση βάσης στοιχείων, εξετάσαμε πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, από ε, εκθέσεις της ε, υπηρεσίας χημικών και κάναμε πάνω από 10 ε, μελέτες. Είναι λοιπόν πλήρως εμπεραστατωμένη αυτή η έκθεση και δείχνει ότι το REACH έχει βελτιώσει σημαντικά την προστασία του περιβάλλοντος ε, και των ανθρώπων, έχει βελτιώσει τις δοκιμές στα ζώα και έχει ε, ε, διασφαλίσει την ομαλή κυκλοφορία των χημικών στην ενιαία αγορά. Προτείνονται 16 συγκεκριμένε δράσει στην έκθεση για να βελτιωθεί η εφαρμογή. Οι τομεί ε, προτεραιότητα που έχουν εντοπιστεί για κατεπίγουσα δράση αφορούν τα κενά στα δεδομένα και στι εγγραφέ, ε, την απλοποίηση τη έγκριση, ε, να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και μη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, να βελτιώσουν τι εφαρμογέ τα κράτη-μέλη, κυρίω για τη βελτίωση τη συνοχή μεταξύ REACH και άλλη νομοθεσία κυρίω ε, τα θέματα προστασία των εργαζομένων και την νομοθεσία περί αποβλήτων. Δύο εδώ επίτροποι, ο Επίτροπο Βέλλα και ο επίτροπο ε, βιομηχανία, η κυρία Μπιανκόφσκα, παρουσίασαν την έκθεση ΡΙΤΣ στα αντίστοιχα Συμβούλια Υπουργών ε, ήδη και συζητιέται περαιτέρω και στις ομάδες εργασίας του Κοινοβουλίου και τα κράτη, το Συμβουλίου συγγνώμη, και τα κράτη-μέλη γενικώ καλωσορίζουν τα συμπεράσματα του ΡΙΤΣ, αλλά παραδέχονται βεβαίω ότι ε, υπάρχει και ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις. Ε, ξεκινάει μια ευρεία συζήτηση με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, με τον Οργανισμό Χημικών και ξέρετε ότι έχουμε αναπτύξει περαιτέρω τις δράσεις που έχουμε προτείνει και προτείνουμε να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με την ε, Υπηρεσία Χημικών και τον κλάδο. Ε, διοργανώνουμε μια διαβούλευση ε, με τους ενδιαφερομένους τον Ιούνιο για να συζητήσουμε περαιτέρω τα θέματα αυτά και να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις 16 δράσεις και καλωσορίζουμε ιδιαίτερα και τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων για να έχουμε και στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ε, ε, καλούμε να συμμετέχετε και στην συνεδρίαση των ενδιαφερομένων. Ενδιαφερόμαστε για τις απόψεις σας τώρα και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις μαζί με τον Κάρλο Πετινέλη για τις απόψεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Ο κύριος Πότσης είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για την παρουσία της εδώ σήμερα. Παρά τον στόχο της ε, διαδικασίας ε, του προγράμματος REACH, όλες οι αιτήσει για την συνέχιση της χρήσης ουσιών μεγάλου ρίσκου έχουν εκχωρηθεί μέχρι τώρα και πάνω από 300 αποφάσεις έχουν υιοθετηθεί μέχρι σήμερα. Υπό το θεματολόγιο τη καλύτερη νομοθεσία του ευνομοθετή, αντί για την προώθηση τη υποκατάσταση αυτών των ουσιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δώσει προτεραιότητα στην ε, απλούστευση και ε, τον εξορθολογισμό αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να, γίνεται, να είναι ακόμα πιο φτηνό και εύκολο για κάποιον να χρήσει και να ε, να χρησιμοποιεί και να παράγει ουσίες υψηλού ρίσκου, περαιτέρω περικόπτοντας το κόστος ε, της υποβολής αίτησης. Ήδη έχει περιοριστεί στο ίμιση το κόστος υποβολής αίτησης το 2013. Με την απλούστευση της διαδικασίας παρέχει μάλιστα κίνητρα για την συνέχιση της χρήσης υψηλού ε, ρίσκου αντί ε, για την υποκατάστασή τους. Και εφόσον δεν έχει απορριφθεί καμία αίτηση, ακόμα και όταν υπάρχουν ξεκάθαρα εναλλακτικέ λύσεις, ε, εμποδίζεται έτσι η ε, διαδικασία του προγράμματος REACH και τη σταδιακής κατάργηση ε, των ουσιών υψηλού κινδύνου. Ε, δεν βοηθάει και την καινοτομία και την χρήση πιο ασφαλών προϊόντων. Τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πετύχει το ΡΙΤΣ, ε, τον βασικό του μέλημα που είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και την προώθηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας με τη σταδιακή κατάργηση των πλέον επικίνδυνων χημικών ουσιών. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξή. Έχω την εντύπωση ότι ήδη έχετε απαντήσει στα περισσότερα από τα ερωτήματά μου. Άκουσα τον ε, προαλήσαντα και πράγματι θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι πιο απλές. Κάποιες φορές μου φαίνεται ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τα πράγματα, για τον κλάδο σε βαθμό που δεν τους ενθαρρύνουμε καν να βρουν υποκατάστατα. Και υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε ένα σύστημα ελεύθερης κυκλοφορίας και διακίνησης των χημικών ουσιών χωρίς κανένα πρόσκομα για τον κλάδο και να μπορεί ο κλάδος να χρησιμοποιεί ε, όλα τα, τα μέσα που θα τους διευκολύνουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό ανεξάρτητα από, τον, από τα επίπεδα ασφαλείας τους. Ένα άλλο ζήτημα τώρα που συνδέεται με την κατάσταση αυτή. Πώς είναι δυνατόν η Ευρώπη να είναι βιώσιμη και να πετύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2020 ε, αν δεν εφαρμόζεται το REACH. Είναι πολύ κακή η εφαρμογή του REACH. Πρέπει εμείς να επέμβουμε σε πολιτικό επίπεδο και να επικεντρωθούμε περισσότερο σε αυτήν μας την προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε τη χρήση του REACH. Νομίζω ότι ε, το πρόγραμμα της καλύτερης νομοθεσίας θα πρέπει να ε, ονομαστεί εκ νέου σε κακή νομοθεσία. Δεν ήταν αυτή η αρχική ε, ουσία του REACH, ο αρχικός στόχος, ε, αλλά δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ευχαριστώ, κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρέμβασή της. Νομίζω ότι το REACH ήταν καλή νομοθεσία για την ε, εξέταση και την έγκριση όλων των χημικών ουσιών με επιβεβαίωσή τους βεβαίως από επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια περίπτωση που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Το πρόβλημα που έχουν οι παραγωγοί αρωματικών φυτών και στη χώρα μου και στη Γαλλία ε, είναι αυτά τα οποία γνωρίζω καλύτερα. Για αυτούς η εφαρμογή της νομοθεσίας REACH ε, η οποία στόχο έχει να προστατεύσει την δημόσια υγεία από την χρήση επικίνδυνων χημικών ε, ουσιών, απαιτεί χημική απόδειξη, επιστημονική απόδειξη ότι όλες οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι υπό έλεγχο. Όλα αυτά αφορούν τα εθέρεα έλαια και σημαίνει ότι χρειάστηκε να εφαρμόσουν πολύ περίπλοκες διαδικασίες ανάλυσης των ουσιών που περιλαμβάνονται στα εθέρεα έλαια ε, λεβάντας ε, και σημαίνει ότι αυτές οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, σχετίζονται και άμεσα με την Ήπεθρο, ε, πρέπει να καταβάλουν πολύ σημαντικά ποσά και ε, η συμμετοχή σε αυτές τις τόσο δαπανερέ διαδικασίες οδήγησε και σε δημιουργία συνεταιρισμών για να αντιμετωπίσουν αυτό το πολύ μεγάλο κόστος. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προβλέψει κάποια εξαίρεση ή κάποιο πιο ήπιο κανόνα για αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σέτομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα ερώτημα έχω για το REACH. Αυτή τη στιγμή ε, επικεντρώνεται περισσότερο στις ουσίες PBT. Persistent, Bioaccumulative and Toxic. Για παράδειγμα, ε, για τις μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού ε, και επεξεργασίας υδάτων ε, έχουν άλλα προβλήματα. Είναι πολύ διαλυτές ουσίες στο νερό και πολύ τοξικές. Είναι δύσκολο για τις επιχείρησεις αυτές να αφαιρέσουν αυτές τις ουσίες από το τελικό πόσιμο νερό. Υπό αυτή την έννοια θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή, Επιτροπή εάν επικεντρώνεται και ασχολείται και με αυτές τις ουσίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλο. Η κυρία Κάντενμπαχ. Uh, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αφαιρέθηκα για μια στιγμή και δεν είμαι βέβαια. Ίσως να το θέξατε αυτό στην εισαγωγή σας. Από όσο γνωρίζω δεν προτείνονται action points για να βελτιωθεί η συμμόρφωση και ποιότητα των πληροφοριών στους φακέλους καταχωρήσεων. Ενώ αυτό είναι σημαντικό εμπόδιο για την εφαρμογή του REACH. Μέχρι τώρα ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι συνεχίζει με την ήπια προσέγγιση με τις βιομηχανίες αυτές με ενημερωτικές επιστολές παρόλες, παρόλη την αύξηση των μη συμμορφώσεων, επιτρέπεται παρόλα αυτά η πρόσβαση στις αγορές, επειδή δεν υφίσταται ε, συνέπειες. Χωρίς τις δράσεις αυτές όμως, θα, συνεχίσει να, θα συνεχίσουν το φέρουν το βαρός οι χώρες μέλη για να συμπληρώνουν τις αναγκαίες προφορίες για ορισμένες διαδικασίες REACH όπως ε, λίστες υποψηφίων κλπ. Εμείς θέλουμε εφαρμογή της αρχής no data, no market. Εφόσον δεν δίνετε δηλαδή τα απαραίτητα δεδομένα, δεν έχετε πρόσβαση στην αγορά. Άλλος κανείς? Κύριε Σαντάσκας, έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστώ. Και πάλι. Θα απαντήσουμε από κοινού, πρώτα εγώ και μετά ο συνάδελφος, για την υποκατάσταση των ουσιών που ήταν το πρώτο ερώτημα. Οφείλω να διαφωνήσω μαζί σας εδώ. Γιατί είμαστε βέβαιοι και το έχουμε διερευνήσει το θέμα. Όταν μια ουσία τίθεται στον κατάλογο των υποψηφίων ουσιών, όχι στον κατάλογο της αδειοδότησης, οι επιχειρήσεις ήδη αρχίζουν, να, ήδη αρχίζουν να επενδύουν ε, στην έρευνα και ανάπτυξη ε, σε ό,τι αφορά την υποκατάσταση. Αυτό είναι βέβαιο και είναι αρκετά πιθανό στις περισσότερες περιπτώσεις όταν τίθεται στην, ε, στον ένα τον άλλο κατάλογο αυτές τις ουσίες, αυτό είναι ήδη ένδειξη ε, προς τις επιχειρήσεις ότι αυτό μπορεί να είναι, δημιουργηθεί πρόβλημα αυτή την ουσία και έτσι τους δίνουμε κίνητρο να εξετάζουν εναλλακτικέ λύσεις. Ε, υπάρχει λοιπόν υποκατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές είναι αρνητική η υποκατάσταση. Ξέρουμε ότι μπορεί να απογορευτεί μια ουσία μέσω του REACH και να χρησιμοποιηθεί μια άλλη ουσία που δεν έχει απογορευτεί ακόμα, όμως έχει αντίστοιχε ιδιότητες και έτσι η υποκατάσταση αυτή δεν μας βοηθάει ουσιαστικά. Αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε νέες προσεγγίσεις, ομαδοποίηση συναφών ουσιών για παράδειγμα και κοινή αντιμετώπιση τους. Ε, διαφωνώ επίσης με την κυρία Άουκεν για την γενικευμένη αποτυχία του REACH. Αυτό είπα στην αρχή, ότι είναι ε, πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία. 17.000 ουσίες έχουν καταχωριστεί μέχρι τώρα και σας διαβεβαιώ ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων χημικών ουσιών στον κόσμο. Μέσα σε μια δεκαετία φτιάξαμε κάτι που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έχουμε την ε, πιο στρατηγική σημασία ε, βάση δεδομένων στον κόσμο. Αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει αποτυχία. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα και προκλήσεις. Αναφέρατε την ποιότητα των φακέλων καταχώρησης. Όντως, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα και δυναμίες ως προς την ποιότητα. Προσπαθούμε να τα επιλύσουμε μαζί με τον αρμόδιο οργανισμό χημικών ουσιών. Ο οργανισμός εξετάζει ακόμα και μία προς μία ε, τις περιπτώσεις καταχώρησης και όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση ε, έρχονται σε επαφή με τον κλάδο και ζητούν την επικαιροποίηση των στοιχείων. Βέβαια, βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα του συστήματος. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν θετικό κλίμα συνεργασίας με τον κλάδο, Όμω και πάλι πρέπει να βρούμε νέα κίνητρα για την ε, επικαιροποίηση των στοιχείων για τι επιχειρήσει. Γιατί κάποιε φορέ οι επιχειρήσεις ε, καταχωρίζουν μια χημική ουσία, μετά υπάρχει όμω εξέλιξη. Ε, αλλάζουν τα πράγματα, νέα χρήση, νέε ποσότητε, νέα επιστημονική γνώση και κάποιε φορές ε, δεν επικαιροποιείται ο φάκελο. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα για την διόρθωση αυτού του προβλήματος, προκειμένου να επικαιροποιούνται η Και μετά είναι και το ζήτημα της αξιολόγησης. Γιατί δεν είναι... Δεν απαιτείται μόνο σωστή καταχώρηση, αλλά και σωστή αξιολόγηση, που είναι αρκετά επαχθής διαδικασία, δαπανηρή. Ε, απαιτείται και, απαιτείται και δοκιμές, ορισμένες φορές και δοκιμές σε, σε ζώα. Είναι κάτι λοιπόν που μας απασχολεί. Γι' αυτό που είπατε λοιπόν για τους φακέλους καταχώρησης, ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση και δεν προτείνουμε κάτι, αν δείτε την υπαριθμόν 1 ενέργεια, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Πώς θα βελτιώσουμε τους φακέλους. Και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερως και είμαστε σε επαφή με τον κλάδο. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Ουσίες στο πόσιμο νερό. Το REACH ισχύει ε, για όλες τις ουσίες ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται, πού μπορούμε να την εντοπίσουμε. Πρέπει όμως να εξετάσουμε τις προβληματικές ιδιότητες των χημικών ουσιών που εντοπίζονται σε διαφορετικούς τομείς, νερό, προϊόντα καταναλωτών κτλ. Μπορούμε εδώ να πούμε ότι έχουμε νέα πρωτοβουλία για το πόσιμο νερό. Πράγματι, προτείνουμε την ε, επίλυση του ζητήματος ε, με αυτές τις προβληματικές ουσίες και έτσι αυτές οι δύο προτάσεις θα κινηθούν από κοινού και το REACH και η πρόταση για το πόσιμο νερό. Να δώσω τώρα το συνάδελφο, με την έλεγχη για να απαντήσει τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να συμπληρώσω την, ερώτηση ε, της κυρίας Σάουκεν. Τα αποτελέσματα της ε, αναθεώρησης του ΡΙΤΣ είναι ε, σαφή έχει συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος και έχει προωθήσει ε, εναλλακτικέ λύσεις στις δοκιμές ε, των ζώων. Επομένως, σε καμία περίπτωση μπορούμε να, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ελλειπής η εφαρμογή του ΡΙΤΣ. Είναι ε, αποτελεσματική, η διαδικασία εφαρμογής του ΡΙΤΣ δεν έχει ολοκληρωθεί και η έκθεση ήδη έχει εντοπίσει 16 τομείς στους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η εφαρμογή. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι μόλις ξεκίνησε το τρίτο στάδιο της εφαρμογής του REACH, ε, διότι ε, το 2018 έχουμε το στάδιο ε, χαμηλή, χαμηλού τονάζ των χημικών προϊόντων, επομένως θα πρέπει να βρουν λίγο τους ρυθμούς τους οι κάποιες βιομηχανίες, αλλά δεν συμφωνούμε με την ερμηνεία σας ότι είναι και πολύ φτωχή η εφαρμογή του REACH. Τώρα, το τρίτο στάδιο για το 2018 μου επιτρέπει να απαντήσω και στην κυρία Γιούζο. Ε, προφανώς ε, και γνωρίζουμε ότι η εφαρμογή ενός κανονισμού, οποιοδήποτε και να είναι, είναι δαπανηρή και υπάρχει κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι να ε, προσφέρουμε εξαιρήσεις. Αυτή είναι η βασική αρχή. Ε, πολλές φορές έχουμε συναντηθεί με τους παραγωγούς εθέρων ελαιών και ε, έχουμε διευκρινίσει ότι δεν μπορούμε να δώσουμε εξαίρεση για τα εφαίρεα έλαια ε, επειδή είναι παραοϊόν γεωργίας ή χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Τα εφαίρεα έλαια ε, θεωρούνται ουσίες οι οποίες ε, προκαλούν κάποια ανησυχία, επομένως πρέπει να χρησιμοποιηθεί το REACH και το αποτέλεσμα είναι ότι ε, επειδή ακριβώς θέλουμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία ε, Χημικών έχει προτείνει κάποια μέτρα για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν προς τον κανονισμό REACH. Υπάρχουν κάποια σεμινάρια. Νομίζω στη Γαλλία υπάρχει και κάποια χρηματική ε, στήριξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φυσικά είμαστε διατεθειμένοι να παρέχουμε και κάτι αντίστοιχο σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε εξαίρεση για ουσίες οι οποίες θεωρούνται ε, ουσίες ε, ανησυχίες γιατί ε, παράγονται από μικρές επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει ανησυχία υπάρχει για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι και ευχαριστώ και τους κυρίους Αντράουσκα και κυρίους Πετινέλη επειδή, που απάντησαν τις ερωτήσεις. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει κάτι τα διάφορα. Επόμενη συνεδρίαση 25 και 26 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Είστε πανίδι.